στήσει τον κύριο Παύλο Ιγκλέσιας. Η κυρία Μαρία Χιμένες Παρμπάτα επίσης εκλέχθη ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ε, αντικαταστήσει τον κύριο Φερνάδο Μπαραντελάν. Και αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Νοεμβρίου 2015. Το Κοινοβούλιο λοιπόν σημειώνει την εκλογή και αναγνωρίζει την εκλογή του κυρίου Μπενίτο Ζιλουάγκα και τη κυρία Χιμένε Μπαρμπάτη. Καλώ ορίζουμε τα νέα μέλη στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι θα συμμετάσχουν στι συναντήσει και συνεδριάσει του Κοινοβουλίου και των σχετικών σωμάτων με πλήρη δικαιώματα και προνόμια όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό. Η GUNGL